σε περίπτωση βέβαια που έχουμε και τα σχετικά στοιχεία από τα κράτη-μέλη για να δώσουμε περισσότερες κατευθύνσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώνουμε εδώ το σημείο αυτού της μεσιάς διάταξης και η ψηφοφορία για την έκθεση αυτή θα γίνει αύριο στις 12.30. Περνάμε στο επόμενο σημείο της μερισιάς διάταξης που είναι και το τελευταίο για απόψε. Έκθεση του συναδέλφου Σουίνμπερν με θέμα ρύθμιση των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα. Αδιαφανείς δεξαμενές, dark pools κτλ. Το λόγο έχει ο κύριος εισηγητής για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να εξηγήσω στους αμύητους τι αφορά η έκθεσή μου. Η έκθεσή μου αφορά συναλλαγή σε χρηματοπιστωτικά μέσα συμπεριλαμβανομένων των ε, dark pools, ε, δηλαδή ανταλλαγές μετοχών που δεν εμφανίζονται πουθενά. Η έκθεση γενικότερα αφορά την εφαρμογή της οδηγίας ε, περί χρηματαγορών του 2007 που αφορά τις χρηματαγορές και τα μετοχικά κεφάλαια. Παρά το ότι είναι πολύ τεχνική η έκθεση, χάρηκα για το επίπεδο της συζήτησης που είχαμε στην Επιτροπή και χαίρομαι για το ότι οι συναδελφοί μου στήριξαν αυτή την έκθεση. Και 194 τροπολογίες έγιναν 26 συμβιβαστικές τροπολογίες, οι οποίες στήριξαν περισσότερες ομάδες. Δεδομένου του χρόνου στον οποίο έρχεται αυτή η έκθεση και το ότι θα ψηφιστεί στην Ολομέλη αυτή την εβδομάδα, θεωρώ πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσθέτει εδώ πέρα στην διαβούλευση της Κομισιόν για την MIFID 2 την οδηγία για τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Ε, ζητάμε εδώ πέρα να ερευνηθούν αυτή τη στιγμή τα μέρη όπου γίνονται αυτές οι συναλλαγές. Κυρία Σούινμπορν, λέει ο πρόεδρος, σας οικετεύω να επιβραδύνετε λίγο γιατί έχουμε πρόβλημα με τους Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει έτσι μια σειρά έρευνών στα σημεία εκείνα όπου γίνονται συναλλαγές και ρυθμίζονται από την σχετική οδηγία έτσι ώστε οι ίδιες υπηρεσίες να ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο. Θεωρώ λοιπόν πως το έγγραφο της Κομισιόν μπορεί να έχει πάει ένα βήμα παραπάνω με το να διευρύνει τον ορισμό του για να μπορούμε εδώ πέρα να καλύψουμε όλες τις αγορές και πωλήσει οπουδήποτε συναντούνται αγοραστές και πολιτές για να κλείσουμε ένα παραθυράκι και εξασφαλίζεται έτσι η αναλογικότητα καθώς υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση εντός των κατηγοριών για MDF, SI, BCN και παράγωγα. για να υπάρξει επιπλέον και μια εξέταση των dark pools, κάτι το οποίο νομίζω θα καλωσορίσουν και οι επενδυτές και ε, καθώς νομίζω πως υπάρχει τουλάχιστον η δυνατότητα κατάχρησης. Οπότε θα πρέπει νομίζω να συνεχίσουν να υπάρχουν για να μπορούν να τις χρησιμοποιούν όσοι θέλουν για να εκτελέσουν παραγγελίες των μετοχών τους χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως γίνεται κατάχρηση αγοράς ή χειραγωγήσει των τιμών. Επίσης, πέραν από τα, τις οδηγίες MIFID, θεωρούμε με την Κομισιόν πως πρέπει να υπάρξει μια αναδιατύπωση και επανορισμός, καθώς η δυνατότητα αυτή τη στιγμή να γίνει αρμπιτράζ μεταξύ των κρατών μελών για να βρεθεί η ευνοϊκότερη ερμηνεία των κανόνων δεν θα πρέπει πλέον να αποτελεί μια δυνατότητα. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης είναι σαφές πως το μεγαλύτερο έλλειμμα εφαρμογής της οδηγίας περί χρηματαγορών είναι το ότι δεν υπάρχει το ότι δεν υπάρχει μία ε, ενιαία ένα ευρωπαϊκό ενοποιημένο δελτίο παρακολούθησης, κάτι το οποίο φαίνεται ακατανόητο στου αμερικανού επενδυτές. Εδώ όμω και τρία χρόνια οι συμμετέχοντε στην αγορά δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν κάτι τέτοιο. Και η Επιτροπή μας λοιπόν δεν θέλει να πάει πέρα από το να δώσουμε εντολή για αυτά τα οποία ορίζει ο Εάν όμως δεν βρει μια λύση η αγορά θα αναγκαστούμε να παρέμβουμε. Βεβαίω όλα αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο έντονη συζήτηση ε, στην ε, αγορά μας για διάφορες ε, καταχρηστικές πρακτικές. Όμως δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε στον ρόλο κάποιων συμμετεχόντων στην αγορά, ιδιαίτερα του εάν είναι εύκολο να... και αν είναι χρήσιμο να υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες αστραπιές και υψηλού όγκου εντολές. Να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο ρόλος του, θετικός ή αρνητικός, πριν προτείνουμε νομοθετική δράση να είμαστε σίγουροι πως έχουμε δεδομένα για να μην επιβάλλουμε νομοθεσία η οποία θα καταστρέψει την αποτελεσματική λειτουργία των ευρωπαϊκών αγορών. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει να δούμε την ακαιρεότητα των αγορών. Οι αγορές δεν είναι μόνο για τους ενδιάμεσους, αλλά για να μπορέσουν οι επενδυτές να δώσουν κεφάλαιο στις επιχειρήσεις για να δράσουν στην πραγματική οικονομία. Αυτή η βασική λειτουργία των αγορών πρέπει να είναι στο νου όλων μας, καθώς θα περάσουμε στην οδηγία MIFID 2. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε κυρία Σουίνμπερν και σας ζητώ συγγνώμη που σας απεκάλεσα κύριο ε, Σουίνμπερν στην αρχή γιατί αυτό έβλεπα μπροστά στο έγγραφο μου. Ζητώ συγγνώμη. Δεν θα το ξανακάνω. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Σας διαβεβαιώ. Και πάλι λοιπόν, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, έχουμε τώρα τη διαδικασία προσέλκυσης της προσοχής του Προέδρου, Catch the Έχουμε τρεις συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο, επειδή ε, η συζήτηση είναι σημαντική και έχουμε και χρόνο στη διάθεσή μας. Θα παραχωρήσω 1,5 λεπτό στον καθέναν από τους ομιλητές. Σας παρακαλώ βέβαια να σεβαστείτε τον 1,5, το 1,5 λεπτό. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Φιλίπ Ζουβά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το κείμενο αυτό είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Περί τίνος πρόκειται. Πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Δεν θα πρέπει τα πράγματα να συνεχίσουν να γίνονται όπως παλιά. Πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Πρέπει να υπάρξει τάξης πλέον στο σύστημα. Αυτοί οι οποίοι σήμερα εποφελούνται στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κρίση και από την αγωνία των πολιτών τα ρίχνουν όλα στην Ευρώπη. Λένε η Ευρώπη φταίει που δεν δουλεύει το σύστημα, το ευρώ φταίει που δεν δουλεύει το σύστημα και να φύγουμε από το ευρώ λένε ορισμένοι. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά για να αποδείξουμε ότι έχουμε ανάγκη από κοινού κανόνες για να αποδείξουμε ότι οι χώρες της Ευρώπης αν δεν ήταν ενωμένε θα είχαν πεθάνει οικονομικά σήμερα. Έχουμε ανάγκη από κοινέ πολιτικές, έχουμε ανάγκη από κοινή λειτουργία και εναρμονισμένη λειτουργία του συστήματος. Είναι απλό το θέμα ουσιαστικά. Από κοινού είμαστε ισχυροί. Μεμονωμένοι είμαστε νεκροί. Ευχαριστώ κύριε Ζουβά. Τσέγγεντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί είστε γενιόδωρος με το χρόνο τον οποίο μας δίδετε. Η έκθεση της κυρίας Σουίνμπερν είναι πάρα πολύ σημαντική σχετικά με τη ρύθμιση των χρηματαγορών. Ποιο είναι το λάθος το οποίο όμως επαναλαμβάνεται. Ζητάει να υπάρξει περισσότερος διακανονισμός. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αργά πια. Ο διακανονισμός και ο έλεγχος μέχρι τώρα ήταν περίπλοκος, μη κατανοητός. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε σωστά αυτά τα οποία έχουν συνέβη και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε τις μεγάλες επενδυτικές προσπάθειες από τις προτάσεις αυτές. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε σωστά και να καταστήσουμε τους κανόνες που υπάρχουν πιο αυστηρούς όπου αυτό είναι δυνατόν. Γιατί τα παράγωγα προϊόντα δημιουργούν μερικές φορές πληθωριστικές τάσεις. και έτσι όπως δουλεύει το σύστημα φοβάμαι ότι οι πλούσιοι θα γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Ευχαριστώ. Τον τελευταίο λόγο στη συζήτηση αυτή θα έχει η αγαπητή συνάδελφος Μπασέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση Swinburne μιλάει για την δημιουργία ίσων όρων σε πολυμερή μέσα συναλλαγών. Θεωρώ πως ε, είναι σημαντικό να δούμε και την ε, επιτήρηση των μέσων αυτών, να περιοριστεί ο συστημικός κίνδυνος και να διασφαλιστούν συνθήκες σωστού ανταγωνισμού. Ανησυχώ πως δεν υπάρχουν εδώ πέρα πληροφορίες για τις στρατηγικές συναλλαγών. Η μόνη δυνατότητα να αντιληφθούμε πράγματι αν η αγορά λειτουργεί σωστά ή όχι είναι μέσω των ε, ρυθμιστικών αρχών από τις οποίες μπορούμε να λάβουμε τις κατάλληλες πληροφορίες. Η υπηρεσία έμζα θα πρέπει να ορίσει κοινούς κανόνες αναφοράς ε, και για τα χρηματιστήρια και βεβαίως για τις συναλλαγές εκτός χρηματιστήριων. Θα ενδιαφερόμουν να ακούσω παραδείγματος χάρη μια αξιολόγηση αντικτύπου για το ε, ελάχιστο ε, ρύθμιση των ανωνύμων πλατφορμών. Έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε μια ελάχιστη ροή πληροφοριών για αυτές τις συναλλαγές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο, στον Επίτροπο Χάν, για να απαντήσει. Και με την παρέμβασή του θα κλείσει το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Κύριε Επίτροπε. Uh, Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Επιτρόπου Μπάνιε θα ήθελα να απαντήσω λέγοντας ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τη διαφάνεια στις χρηματαγορές και όλοι οι τομείς που συναποτελούν τις αγορές θα πρέπει να υπόκεινται σε σωστό έλεγχο σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας των 20. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Εμείς ξέρετε ότι έχουμε περάσει σε έναν έλεγχο τώρα πλέον ε, της αγοράς των παραγόγων οι συστάσεις ε, τις οποίες κάνετε είναι ενσωματωμένες θα έλεγα στις σκέψεις τις οποίες κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δημοσιεύσει το 2011. Η αναθεώρηση του ΜΙΦΕΔ νομίζω ότι θα βοηθήσει το σύστημα να λειτουργήσει καλύτερα για την κοινωνία και την οικονομία. Νομίζω ότι από τον επόμενο μήνα που θα τεθούν σε ισχύ και οι νέοι εποπτικοί μηχανισμοί, οι νέες εποπτικές αρχές ε, τα πράγματα θα βελτιωθούν. Ζητάμε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε να περάσουμε ταχύτατα τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα. Το ΜΥΦΕΝΤ είναι ο θεμέλιος λίθος του νέου διακανονιστικού πλαισίου των χρηματαγορών είναι κάτι το οποίο προϋπήρχε της χρηματοπιστωτικής κρίσης αλλά παρόλα αυτά διευκόλυνε τα πράγματα να εξελιχθούν ομαλά ακόμα και μετά τις τελευταίες δυσκολίες. Προφανώς και υπάρχουν κάποια προβλήματα. Οι τεχνολογικές αλλαγές στις χρηματαγορές διασφαλίζουν έτσι ώστε οι διακανονιστικές ρυθμίσεις οι οποίες ήταν ενήμερες και επίκαιρες πριν μερικά χρόνια να μην είναι πλέον σήμερα και γι' αυτό ακριβώς στα πλαίσια της διαβούλευσης που ξεκινάμε θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι αναγνωρίζοντας ότι οι βασικοί στόχοι του ΜΙΦΕΔ εξακολουθούν να είναι σωστοί και έγκυροι και το θέμα είναι να διασφαλίσουμε τις χρηματαγορές, να κρατήσουμε ανοιχτές τις επενδυτικές δραστηριότητες και να διασφαλίσουμε επίσης και τους επενδυτές γενικά ανοιχτές τις πόρτες των χρηματαγορών. Υπάρχει ανάγκη για βελτίωση σε πολλούς τομείς ε, ε, των χρηματαγορών, ιδιαίτερα των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ισότιμη συμμετοχή και δυνατότητα των επενδυτών. Πρέπει να βελτιώσουμε επίσης τους κανόνες της διαφάνειας οι οποίοι εφαρμόζονται σε όσους συμμετέχουν στις χρηματαγορές. Ένας άλλος σημαντικός τομέας από την κυρία Σουίνμπερν είναι η βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς των παραγόγων σύμφωνα με τις αρχές της ομάδας των 20. Ταυτόχρονα πρέπει να βελτιώσουμε τους υπάρχοντες κανόνες σχετικά με την προστασία των επενδυτών διασφαλίζοντας ότι όλες οι πρακτικές καλύπτονται από τους ισχύοντες κανόνες είναι βασικό συστατικό για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του επενδυτή. Λοιπόν, οι νέες μορφές εποπτείας ε, νομίζω θα βελτιώσουν τη λειτουργία των χρηματαγορών. Έχω την αίσθηση ότι έτσι θα μπορέσουν να δουλέψουν καλύτερα οι νέες αγορές μετοχών ε, και επενδυτικών μέσων. Είμαστε σε επαφή, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και με τις Ηνωμένε Πολιτείε για να διασφαλίσουμε τη διεθνή σύγκληση και ε, κάποιες τρευλώσεις του ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο τομέα. Η έκθεση Swinburne νομίζω ότι έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις αλλαγές στον διακανονισμό των αγορών. Οι αναλύσεις σας και οι συστάσεις σας συμπίπτουν εν πολλής με τις δικές μας.